Επιτροπής. Δίνω το λόγο εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κυρία Τάισεν. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Πρόεδρε, εξαιρετικοί κυρίε και κύριοι, με χαρά έρχομαι να σας παρουσιάσω την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για στοχευμένε τροποποίησει στην ε, οδηγία για την απασπάση των εργαζομένων που υιοθέτησε ο συλλογικό όργανο η Επιτροπή σήμερα εδώ στο Στρασβούργο και θέλω να σα πω ότι είναι ακόμα νοπό το μελάνι τη πρόταση. Η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών είναι δύο από τι τέσσερι θεμελιώδεις ελευθερίε τη εσωτερική μα αγορά, Από την ανάληψη των καθηκόντων μου δεν άκουσα κανεί να αμφισβητεί αυτέ τι θεμελιώδει ελευθερίε, αλλά άκουσα συχνά να εκφράζονται ανησυχίε για τέσσερι συγκεκριμένε πτυχέ αυτών. Πρώτον, κινητικότητα ω προ τι χώρε και προελεύσεω και υποδοχή. Δεύτερον, πραγματική υλοποίηση των υφισταμένων κανόνων. Τέταρτον, ε, τρίτον, ε, συγκεκριμένη ισορρόπηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Πολλέ φορέ θεωρείται ότι είναι αθέμητη και ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι δεν πρέπει τις ανησυχίε αυτές να τι αγνοήσουμε, πρέπει να δώσουμε απάντηση σε αυτές. Ποια θα είναι λοιπόν τα κύρια στοιχεία της απάντησής μας, της ανταπόκρισής μας. Θα σας πω ότι καταρχάς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε αντί των ευθυνών, ε, θα υπερασπιστούμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε και μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα ο πολίτης, η αγορά εργασίας και η κοινωνία γενικότερα να υποφεληθούν από τις εξελίξεις. Δεύτερον, χρειαζόμαστε κανόνες σαφείς, δίκαιους και τηρούμενους κάθε φορά στο σημείο πρέπει να τηρούνται και σε αυτό δεν έχουμε επιτύχει πολλά, χρειάζεται ακόμη βελτίωση. Θεωρώ ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία ήδη που επιτρέπουν στις αρχές να εξασφαλίσουν την ελεύθερη διακίνηση σε όρους δίκαιους και αυτή είναι το Γιούρις, αυτά τα εργαλεία είναι το Γιούρις, η πλατφόρμα για την καταπολέμηση της μη δηλωμένης εργασίας, την οδηγία για την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων και την εφαρμοστική οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Αυτά τα τέσσερα λοιπόν εργαλεία θα πρέπει ε, να υλοποιούνται, εφαρμόζονται αμέσως και παρέχουν οι υπηρεσίες μας βοήθεια προς τα κράτη-μέλη από τη στιγμή όμως που έχουν περάσει οι προθεσμίες για την μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο των Σχετικών Οδικιών, τον Ιούνιο δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας εμβεβαιώ δεν πρόκειται να διστάσει να επιβάλλει και μέτρα επιβολής. Μια ελεύθερη αγορά εργασίας θα υπάρξει μόνο εάν τηρούνται πάντοτε και οι κανόνες που έχουμε ε, εγκρίνει εφαρμογή των κανόνων λοιπόν. Ένα κομμάτι όμως της απάντησης μόνο. Και για να προχωρήσουμε πρέπει να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο, να επικαιροποιήσουμε και να ενισχύσουμε τους κανόνες όπου αυτό χρειάζεται. Με το στόχο αυτό λοιπόν ολοκληρώνουμε και την ε, πρόταση, ολοκληρώσαμε στα τέλος του 2015 την ε, πρόταση για την διακίνηση των εργαζομένων, αλλά ξέρετε ότι αποφασίστηκε να αναβληθεί ω ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ρυθμιστεί πρώτα το ζήτημα του Ηνωμένου Βασιλείου και να μην ε, υπάρξει παρεμβολή σε σχέση με συνεχιζόμενε πολιτικέ συνομιλίε. Τώρα που υπάρχει επιτάπητο αυτή η πρόταση για το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε την πρότασή μα για την αναθεώρηση των κανόνων ε, συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης μέχρι ότου βγουν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο αλλά υπάρχουν άλλα ζητήματα κοινωνικότητας και απόσπασης όπου μπορούμε να προχωρήσουμε και σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αθέτει την νομοθετική πρόταση που είχαμε προεξαγγείλει και μέσα στο πρόγραμμα του 2016. Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφή για την πολιτική μου τοποθέτηση. Χρειάζεται περισσότερη απόσπαση εργαζομένων και όχι λιγότερη στην Ευρώπη. 1,9 ε, εκατομμύρια θέσει απόσπαση υπάρχουν. αυξανόμενε τάσεις μεν, αλλά παραμένει ε, λιγότερο από 1% του εργατικού μα δυναμικού αυτό. Χρειάζεται, υπάρχει λοιπόν περιθώριο για ακόμη περισσότερο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πιέσει ώστε να ε, αποδιαρθρωθούν οι φραγμοί ως προς τις εσωτερικές διατάξεις ε, πέραν των συνόρων για αποσπάσεις. Αλλά ταυτόχρονα αυτό θα γίνει με ένα σύστημα οργανωμένο κατά τρόπο θεμητό, ισότιμο για τον εργαζόμενο αλλά και για τις επιχειρήσεις. Πολλά υπόθηκαν, πολλά γράφτηκαν για τη διάρθρωση μεταξύ των κανόνων της ιστορικής αγοράς και των κοινωνικών κανόνων στην Ευρώπη. Για ορισμένου θα πρέπει να επικρατούν οι κανόνε τη ελεύθερη αγορά, για άλλου περισσότερο η κοινωνική προστασία. Ωστόσο, κατ' ουσίαν, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο σημαίνει ότι και τα δύο αυτά σκέλη μπορούν να προχωρήσουν παράλληλα. Και αυτό ήταν ο κύριος στόχος της ε, οδηγίας για την απόσπαση του 1996. Παραμένει δε στόχος της σημερινή μας προτάσεως. Θέλουμε να προαγάγουμε τις υπερσυνοριακές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την προστασία του εργαζομένου και ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των τοπικών και υπερσυνοριακών παρόχων υπηρεσιών στα 20 χρόνια από την υιοθέτηση της οδηγίας του 1996. Η ευρωπαϊκή αγορά εργασία βεβαίως έχει αλλάξει. 28 κράτη-μέλη πλέον. Και οι αποκλήσει σε συστήματα εργασιακά αλλά και μισθολογικά μεταξύ των κρατών μελών ε, είναι όλο και μεγαλύτερες Αντί για περισσότερη σύγκληση βλέπουμε μεγαλύτερες αποκλήσει. και αυτό βέβαια έχει συνέπειες και προς την απόσπαση. Τα χάσματα στους ελάχιστου μισθού έχουν περάσει από ένα λόγο ένα, του ενός τρίτου στο 1 προς 10 από το 1996 το 2016 και όλα αυτά τα οποία αποτελούν στατικά στοιχεία της αμοιβή στην κάθε χώρα έχουν επίσης αλλάξει. Ένα εργαζόμενο μπορεί να έχει 13ο μισθό, μπορεί να έχει δώρο Χριστουγέννων, μπορεί να έχει συνθήκε εργασία ε, σχετικέ με το ταξίδι, χρόνο ανάπαυση για λόγου ε, ταξιδιού. Όλα αυτά δεν καλύπτονται στην οδηγία για την απόσπαση και άρα υπάρχει βεβαιότητα και προβλήματα σε καθημερινή βάση. Πράγμα κακό για τον εργαζόμενο, ο οποίο μπορεί να μην εξασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων του, αλλά και για την επιχείρηση που θα χρησιμοποιήσει τον αποσπόμενο εργαζόμενο, γιατί το κόστος των συναλλαγών είναι πολύ υψηλό και πολλές επιχειρήσεις εγκαταλείπουν ακόμη και την ιδέα της απόσπασης γιατί θεωρούν υπερβολικά περίπλοκη. Σε μια άκρος ανταγωνιστική εσωτερική αγορά, ο ανταγωνισμός στηρίζεται στην ποιότητα, την παραγωγικότητα, την καινοτομία. Το εργασιακό κόστος είναι ένα μόνο στοιχείο αυτών. Αλλά δεν μπορεί ο ανταγωνισμός να στηρίζεται μόνο στο κόστο το εργασιακό. Γιατί αυτό δεν είναι προς όφελος του εργαζομένου, το τη επιχείρηση του και της ανταγωνιστικότητα γενικότερα τη Ευρώπη σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, στον χώρο τη οικοδομή, που έχει ακόμα ένα 43% ποσοστό των αποσπάσεων. Δεν περιορίζεται μόνο αποσπάσεις μόνο σε αυτόν και σε άλλου τομεί. δημοσιογράφοι, τραπεζικοί, ε, υπηρεσίες υγείας, ιατροφαρμακευτικό προσωπικό, ε, ιατρικό και νοφιτισλευτικό προσωπικό καλύτερα. Είναι ε, εργαζόμενοι που ακολουθούν το δρόμο τη απόσπασης και χρειάζεται να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους. Και είναι όλο και πιο έντονο το σύστημα της υπεργολαβίας στην αγορά εργασίας που βεβαίως μπορεί να εξασφαλίσει περισσότερη πρόσβαση σε εξειδικευμένε, ικανότητες, δεξιότητες και περισσότερη αποτελεσματικότητα αλλά ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώση τη αγοράς εάν οι επιχειρήσει υπεργολαβίας δεν, δεν υπάρχουν στου ίδιους κανόνες για τι αμοιβέ. Και αν ε, μόνο η μείωση του κόστους οδηγεί στην εξωτερική ανάθεση του outsourcing, τότε μόνο υποβάθμιση και προς τα κάτω σύγκληση και όχι προς τα άνω μπορούμε να έχουμε. Δεν είναι αυτή η εσωτερική αγορά που θέλουμε και δεν είναι αυτή η εσωτερική αγορά που έχουμε προσχεθεί στους πολίτες μας. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε μια στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση του 1996 για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά πρέπει να επικαιροποιηθούν οι κανόνες ώστε να συμμορφωθούν στα τωρινά δεδομένα και θα σας θυμίσω τις δυσκολίες και τις οδηγίες για την επιβολή των διτάξεων. Τα θυμάμαι και ως Ευρωβουλευτή στην εποχή εκείνη στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω όμως ακράδαντα και ειλικρινά ότι μπορούμε πλέον να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα, καθήκοντα κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη προσοχή αφού γράστηκα τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, των κρατών μελών, των εμπλεκομένων φορέων, και ομάδων συμφερόντων και σημειώνω ιδιαίτερα ότι χρειάζεται καλύτερη προστασία για τους αποσπασμένους εργαζομένους, ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων υπηρεσιών εσωτερικών, εγχωρίων και εξωτερικών, περισσότερη ασφάλεια δικαίου, σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας και της αποφυγής των διακρίσεων και βέβαια σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας και των εθνικών συστημάτων προσδορισμού των μισθών. Η πρόταση που υιοθέτησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει απάντηση σε όλες αυτές τις, ε, σε αυτούς στόχους κατά τρόπο ισορροπημένο για τις διατάξεις παραδείγματι για την ε, αμοιβή με βάση και πρόσφατες αποφάσεις του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και με απόλυτο σεβασμό των διατεραιοτήτων σε εθνικό επίπεδο γιατί θα είναι πλέον ε, ελάχιστος μισθός αλλά θα μπορεί να διεκδικηθεί κάθε επίπεδο μισθολογικό στη χώρα απόσπασης. Επίσης οι κανόνες για την κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να υπηρετούν και βέβαια την κοινωνική πρόνοια αλλά και το εργατικό δίκαιο. Και έτσι κάποιο ο οποίο θα είναι προσπασμένο για περισσότερο από 24 μήνε θα θεωρείται ότι έχει ενταχθεί στην αγορά εργασία τη χώρα υποδοχή θα υπάρξει καλύτερη ευθυγράμμιση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων με την οδηγία για την προσωρινή εργασία από υπηρεσίες ανάθεσης ή από υπηρεσίες απασχόλησης που θα ισχύει και για τους αποσπόμενους εργαζομένους. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, ελπίζω ότι θα μελετήσετε την πρότασή μας, την επίσημη, όχι ανεπίσημες που είδα να σχολιάζονται στον τύπο τις τελευταίες μέρες. Ελπίζω ότι θα μελετήσετε λοιπόν την πρότασή μας με πνεύμα ανοιχτό και επικοδομητικό βλέμμα. Όπως γνωρίζετε, είμαι ζητηθμένη να επανέλθω στο Κοινοβούλιο για να συζητήσω ανα πάσα στιγμή τα θέματα αυτά. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται επικοδομητικά με τους συνομοθέτες, προφανώς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με χαρά, με στόχο να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Κάζα. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο Τάισον διότι Πραγματικά έτσι αισθάνομαι. Την ανάγκη να την ευχαριστήσω γιατί επέδειξε τόλμη. Όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την οδηγία αυτή που απέχει πολύ από την τελειότητα, εμείς στο ΕΛΚ πιστεύαμε ότι πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Προφανώς διαφωνίες θα υπάρχουν και δεν θα συμφωνήσουμε όλοι. Ε, αλλά και μέσα στη δική μας την ομάδα είχαμε μακροσκελείς συζητήσεις και δεν ήταν εύκολο για το ΕΛΚ να καταλήξει σε συμφωνία όπως αυτή που έχετε στα χέρια σας σήμερα για αυτή τη νέα πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς η έκκλησή μου σήμερα είναι προς τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Δεν μπορούμε να είμαστε λαϊκιστές σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Το Κοινοβούλιο πρέπει να βεβαιωθεί και να αποστείλει το μήνυμα ότι είμαστε ενωμένοι, ότι ε, θέλουμε να υπάρξει συμβαστική λύση και μαζί με την εισηγήτρια θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πετύχουμε και οι συντονιστέ και οι υπόλοιποι σκιώδει όλων των πολιτικών ομάδων να εγκρίνουν αυτή την πρόταση. Εδώ έχουμε μία βάση για να καταλήξουμε πραγματικά σε συμβαστική λύση. Εάν τα καταφέρουμε, πραγματικά θα αποστείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προ το Συμβούλιο. Διότι το Συμβούλιο και αυτό χρειάζεται να ε, προχωρήσει. Ευχαριστούμε, αλλά υπάρχει γαλάζια κάρτα για σας. Το δέχεστε. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Μίλησατε για τους εκπροσώπους των διαφορών πολιτικών ομάδων. Και θεώρησα ότι οφείλω να διατυπώσω ερώτηση, μια και αναφερθήκατε στις πολιτικές ομάδες. Όταν λέτε ότι θα πρέπει να καταβάλλεται ένας ελάχιστος μισθός. Ε, πώς το εννοείται ακριβώς. κύριο Κάζα, για να απαντήσει. Πράγματι. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι δεν θα κερδίσουν όλοι αυτό ακριβώς που αρχικά ήθελαν. Όμως με αυτή τη διευθέτηση που τώρα έχουμε αυτή τη διαδικασία πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα δούνε και λαβίν ε, μεταξύ των ε, διαφόρων συμφερόντων. Το θέμα δεν είναι τι θέλω εγώ εγωιστικά, τι εγώ εγωιστικά θέλω να πετύχω, αλλά τι μπορώ να ε, εγκαταλείψω από τα δικά μου θέλω για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Εδώ, ε, εάν παραμείνουμε λαϊκιστές, δήμαγωγοι, θα χάσουμε εν τέλει και εμείς. Οι εργαζόμενοι μας ενδιαφέρουν και αυτούς θέλουμε να προστατεύσουμε και τα δικαιώματά τους. Ευχαριστούμε. Στάινρουκ. λεπτά. Um- δεν μας ενδιαφέρει να περιορίσουμε την απόσπαση, αλλά να την διατυπώσουμε κατά τρόπους ισότιμους και δίκαιους μέσα στην Ευρώπη και χαίρομαι κυρία Τάισεν που διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως η εφαρμοστική οδηγία δεν αρκεί μόνη της και ότι πρέπει να μπούμε στη βασική οδηγία. Οι πιέσει των συνδικαλιστικών σωματιτών και ημών των Σολυμοκρατών οδήγησαν και στη βελτίωση των προτάσεων του σχεδίου προτάσεων της προηγούμενης εβδομάδας. Θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίρνει πιο πολύ στα σοβαρά τον κοινωνικό διάλογο. Ίσως μισθός για την ίση εργασία στον ίδιο τόπο είναι αρχή που πρέπει όλοι να σέβονται και οι εργοδότες και αυτό σημαίνει και συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ε, οι ελάχιστες προδιαγραφές δεν μπορούν να θεωρείται ότι αντικαθιστούν τις μέγιστες προδιαγραφές και δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν όλο και λιγότερες ε, ε, διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων. Δεν μπορεί να υποβαθμίσει την προστασία των εργαζομένων. Πρέπει να έχουμε λοιπόν καλές λύσεις έχουν εντωμεταξύ περάσει 24 μήνες όπου επαληθεύεται η ανεπάρκεια του συστήματος στο ίμιση των αποσπασμένων εργαζομένων ε, στον οικοδομικό κλάδο λιγότερο από 6 μήνες εργάζονται άρα δεν μπορούμε να έχουμε 24 μήνες ως κριτήριο για τις, ε, την ισότιμη επασχόληση πρέπει να έχουμε μικρότερο όριο, εξάμεινο ίσως. Επίσης η αλυσιδωτή απόσπαση χωρίς πραγματική ε, ευθύνη με εταιρείε γραμματοκιβώτια ε, ανώνυμες με συνθήκες ε, παραβίασης των εργασιακών και κοινωνικών συνθήκων ολοκληρωμιλότερες παροχές κοινωνικής πρόνοιας όλα αυτά πρέπει η οδηγία για την απόσπαση να τα επανεξετάσει και βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει με συντονισμό και του κοινωνικού συστήματος Ευχαριστώ πολύ Δέχεστε μια μπλε κάρτα του κύριου Σούλτσε Κύριε Στάνιροκ, και εσείς Γερμανίδα είσαστε όπως και εγώ. Μιλήσατε για ίσο μισθό, για την ίση εργασία στον ίδιο τόπο εργασία. Πώς θεωρείστε λοιπόν αυτό για τη Γερμανία συγκεκριμένα. Ίδιος τόπος εργασίας στη Γερμανία τι σημαίνει. Η ίδια περιφέρεια, το ίδιο Bundesland, το ίδιο κρατήδιο, ολόκληρη η επικράτεια της Μοσπονδιακής Δημοκρατίας. Πώς το βλέπετε αυτό στη Γερμανία. Παρακαλώ. Κύριε Στάινρουκ. Χωρίς μικρόφωνο. Ακριβώς αυτό είναι το αίτημά μου. Όλες οι περιφερειακές και τομεακές συλλογικές συμβάσεις και η ελάχιστη μισθή πρέπει να αποτελούν τη βάση αυτής της οδηγίας για την απόσπαση. Γιατί εάν δουλεύουν δύο άνθρωποι στον ίδιο τόπο και κάνουν την ίδια δουλειά, προσφέρουν το ίδιο έργο, τότε πρέπει να υπάρχει και η ίδια αμοιβή και οι ίδιες κοινωνικές παροχές. Είναι νομίζω Μόνο δίκαιο αυτό. Καλώς η κυρία Μάκιντάρ ένα λεπτό. We've just been speaking about... Μιλάμε για την ε, νομοθεσία στο Κοινοβουλίο, αλλά πρέπει να πω ότι δεν είναι καλό παράδειγμα. Είναι το αντίθετο της καλής νομοθεσίας. Είναι κακή ιδέα να ξανανοίξουμε αυτό το φάκελο, ενώ περιμένουμε ακόμα την εφαρμογή της ε, οδηγίας ε, περί επιβολή στα κράτη-μέλη. Ξέρω πως είναι μια στοχευμένη διάταξη, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευπρόσδεκτο για μένα. Όσον αφορά τι λεπτομέρειε, η αρχή τη αμοιβή ε, για την προστασία του εργαζόμενου είναι πολύ ευρύτερη από την αρχική ε, οδηγία που αναφέρεται στην αμοιβή η... αυτό θα έχει μάλλον αντίθετο αποτέλεσμα γιατί μάλλον αρνητικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ενώ η πρόταση δεν αναφέρεται άμεσα στην ίση αμοιβή για ίση εργασία στην ίδια, στο ίδιο σημείο, υποψιάζομαι πως είναι μια απόπειρα από πλευρά της Κομισιόν να προχωρήσει με αυτή την φιλοδοξία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην δημιουργήσουμε άλλη μια νομοθεσία που θα έχει τις μη επιθυμητές συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ. Δέχεστε γαλάζια κάρτα από το συνάδελφό σας στα αριστερά σας. Τον κύριο Έικερ. She said no. Well... Όχι. Είπατε όχι. Ε, καλά. Θα τα βρείτε μετά από τη συνεδρίαση. Η κυρία Ντλαμπαγιώβα, δύο λεπτά. Νομίζω πως κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να μην δεχτεί τη γαλάζια κάρτα και δεν μπορείτε να την ε, αποκαλείτε ε, ε, φοβητσιάρα. Δεν, μπορούν να, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τέτοια φρασεολογία μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Κυρία Δλαμπαγιώβα, κυρία ε, Επίτροπε, αυτή η πρότασή σας για την απόσπαση των εργαζομένων ήταν μεγάλη έκπληξη για μας. Ήδη αυτό αντιμετωπίζεται στη, μέσω της ισχύωσας ε, νομοθεσίας και υπήρχε μια ισορροπία όσον αφορά την μετακίνηση και την προστασία των εργαζομένων και τις ίσες αμοιβέ. Θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο στόχος της αναθεώρησης αυτής της οδηγίας, αν και δεν έχουμε δει να λειτουργεί αρκετά η ισχύουσα νομοθεσία και δεν ξέρουμε ποια θα είναι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτή. Δεν είναι αυτό αντίθετο με την αρχή της καλύτερης νομοθεσίας. Η Επιτροπή ελπίζει πως θα έχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και καλύτερες συνθήκες αμοιβών ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, το πιστεύετε αυτό, δεν ανησυχείτε ότι η ανταγωνιστικότητα των εταιριών από χώρε λιγότερο ανεπτυγμένε θα είναι χειρότερη, ιδιαίτερα όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων. Έχετε δει την πραγματική οικονομία στα κατημέλη συμπεριλαμβανομένων των διαφορών Στι αμοιβέ στα κράτη-μέλη, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Εγώ πιστεύω πως αυτό θα οδηγήσει σε διαμάχε και θα αυξήσει του τους στην κινητικότητα. Δεν έχει οριστεί ε, δεν έχει οριστεί στα κρατημέλη και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διασυνοριακή οικονομία και στις μικρές επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι ανταγωνιστική δεν θα τα βγάλει πέρα ε, παγκοσμίω και περισσότερο χρειαζόμαστε την ανταγωνιστικότητα. Η Άλντε θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Handel. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει πάρει εκρηκτικέ διαστάσει η απόσπαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν κακό αυτό εάν δεν, υπήρχαν, δεν υπήρχε εκρηκτική ανάπτυξη και στι ε, αναφορέ για καταχρήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να περιορίσει τις ε, καταχρήσεις. Ο κύριος Γιουνκέρ μίλησε για ίση αμοιβή, για ίση εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας. Διαβάζοντας την έκθεση μπορώ να διαπιστώσω ότι αυτά τα οποία περιλαμβάνει δεν μιλούν για ίσο μισθό, για ίση εργασία στον ίδιο τόπο εργασίας. Εάν πάρουμε λοιπόν την, ε, ε, το όρο των 24 μηνών ε, για την εξίσωση του απεσπασμένου με εγχώριο εργαζομένο δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα. Ούτε έχουμε λύσει το πρόβλημα για την υποχρέωση, για την ευθύνη του ε, εργοδότη στις αλυσιδωτές αποσπάσεις. Δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα της απόσπασης από το ένα κράτος ε, του εργαζομένου που δεν είναι πραγματικά εργαζόμενος. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ε, κατάχρησης μέσω της δανειζόμενης εργασίας και πάνω απ' όλα δεν έχουμε επιλύσει το πρόβλημα της, του αποτελεσματικού ελέγχου των κρατών μελών για την απόσπαση γιατί η ανταλλαγή πληροφοριών δεν έχει ρυθμιστεί ικανοποιητικά μεταξύ των κρατών. Και κυρία Επίτροπε, δεν αρκούν όλα αυτά. Χρειάζεται ακόμη περισσότερη βελτίωση. Εάν δεν καταθέσει κάτι καλύτερο η Επιτροπή, πρέπει πλέον το Κοινοβούλιο να επιβάλλει ίσο μισθό για ίση εργασία στον ίδιο τόπο εργασία. Ευχαριστώ. Λάμπερτ. Ένα λεπτό και τριάντα δεύτερα. Thank you, President. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή για την παρουσίαση. Νομίζω πως όλοι κατανοούμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλή προστασία των εργαζομένων από όπου και προέρχονται και όπου και αν και ότι δεν θα πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και οι εταιρείε τους λειτουργούν εντός ε, των ε, νομίμων πλαισίων. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός ώστε να ασκηθεί πίεση προς τα κάτω στις αμοιβέ και στις προδιαγραφές και γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανησυχία για τους αποσπασμένου εργαζόμενους σε διάφορους τομεί. Ε, αναγνωρίζουμε ότι η οδηγία για την εφαρμογή θα πρέπει ακόμα να μεταγραφεί σε όλα τα κρατημέλη και ανησυχούμε γιατί αρκετά κρατημέλη δεν έχουν ε, του κατάλληλους πόρους όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας ώστε να είναι πλήρως ε, αποτελεσματικά. Ορισμένοι μας ε, δεν έχουμε πιστεί για την αποτελεσματικότητα ε, θέλουμε να γνωρίζουμε αν περιορισμένη φύση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που συμπεριλαμβάνονται εδώ αν είναι ευθυγραμμισμένη με ε, το 10, αν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο, ε, αν θα πρέπει να δούμε τομεακές και εταιρικέ συμφωνίες και αν όχι γιατί. Όσον αφορά τα πακέτα αμοιβών, φαίνεται ότι είναι καλύτερο από το να καλύπτεται απλά ή αμοιβή, ειδικά όταν βλέπουμε τόσα πολλά απλά η αμοιβή, ειδικά όταν βλέπουμε τόσο πολλά κράτη που ισχύουν τα ελάχιστη, ελάχιστη μισθή, αλλά όχι μισθή επιβίωσης. Η μείωση των αμοιβών δεν είναι ελκυστική φυσικά για τους εργαζόμενους. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα, μπορέ... ότι θα ισχύσουν όλα αυτά για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που έχουμε. Ευχαριστώ. Η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων επιτρέπει τη εταιρεία να στείλουν σαν πακέτο του εργαζομένου σε ξένη χώρα, ενώ υπάρχουν ακόμη άνεργοι που αναζητούν απελπισμένα μία δουλειά. Η εκμίστοση ανθρώπων ξεκινάει από το 2009 και είναι άμεσο αποτέλεσμα τη αρχή αυτή τη νομοθετική πρόταση. Και είναι μια τεράστια προσπάθεια στο να δημιουργηθεί ένα υπερκράτο χωρί να δίνεται σημασία στα εθνικά σύνορα ή τα πρότυπα διαβίωση, κάτι που ε, θυμώνει του ανθρώπου ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ πολλέ φορέ οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν καν να πληρώσουν τη στέγασή του, τη στέγα για τις η εταιρεία τους. Οι ε, ψηφοφόροι μου όμω στην εκλογική μου περιφέρεια έχουν ακόμη λογαριασμού που πρέπει να πληρώσουν και πολλέ φορέ είναι άνεργοι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα αυτών των οδηγιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Μειώνει τα πρότυπα διαβίωση για όλου του Ευρωπαίου μετερίε που πληρώνουν ε, του ελάχιστου μισθού και ένα κύμα οικονομική μετανάστευση που ουσιαστικά ε, συμπιέζει προ τα κάτω του μισθού. Γίνεται λοιπόν, λένε και σαφέστερο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλει να κάνει χοντρά λεφτά. Εδώ ο στόχο είναι να συμπιεστούν τοπικά οι μισθοί. Και βεβαίω αυτό θα μα οδηγήσει σε κατάρρευση. Ε, διότι ε, στι 23 Ιουνίου ο κάθε εργαζόμενο που θα έχει χάσει τη δουλειά του που θα είναι ανεργός με τις πόρτες ανοιχτές προς την ε, μετανάστευση θα πρέπει να πει επιτέλους τη γνώμη του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φτιαγμένη για μια ελίτ των λίγων, όμως οι πολλοί τελικά θα υποβέλουν τη δική τους άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γιασλοβιέφκα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ συνάδελφοι, πρέπει να πω ότι ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο πρώτα απ' όλα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα της ε, απασχόλησης και των κοινωνικών μας ε, προτύπων. Εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, ιδίω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει αυτήν την κοπή απόφαση να αναθεωρήσει την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Σε λιγότερο από δύο χρόνια, μάλλον μόλι πριν από δύο χρόνια και με πολύ δύσκολε διαπραγματεύσει, όλε οι πολιτικέ ομάδε αλλά και όλα τα κατημέλη μελη δέχτηκαν την οδηγία ε, για την εκτέλεση των ε, ρυθμίσεων σε σχέση με την απόσπαση των εργαζομένων προσωπικώ, θεωρώ ότι είναι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντί να καταμετρήσει τι συνέπειε τη οδηγία για την εφαρμογή τη νομοθεσία αυτή, δεν άκουσε τι είπαν τα κράτη-μέλη και θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία ε, γιατί το ζητούν κάποια κράτη-μέλη. Εδώ όμω αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι ίσω ανταγωνισμό για όλε τι επιχειρήσει. Σίγουρα αυτό ευαγγελιζόμαστε. Όμω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να θυμηθεί ότι οι εταιρείε που υποχρεώνουν τους εργασμένους τους σε απόσπαση ουσιαστικά προκαλούν μεγαλύτερο κόστος για τις επιχειρήσεις ε, σε τοπικό επίπεδο, εκεί όπου αποσπώνται οι εργαζόμενοι. Αυτό λοιπόν να δημιουργεί θέμα των ανταγωνισμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι πολλέ φορέ, εργάζονται και κερδίζουν τους μισθούς τους εις βάρος των τοπικών αγορών. Όμως η απόσπαση αφορά σε μεγάλο βαθμό την Ανατολική Ευρώπη από που μετακινούνται εργαζόμενοι προς τη Δυτική. Εδώ λοιπόν μπορεί να δημιουργηθούν γκρίζε ζώνες και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει από την άποψη των κοινωνικών μας συστημάτων της κοινωνικής πρόνοιας. Ελπίζω ότι χάρη δουλειά, στην δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορέσουμε να φτάσουμε ο πρόεδρος διακόπτη, ο κύριος, η κυρία για δύο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, το περασμένο Σαββατοκύριακο η δική μου χώρα ε, είδε πρώτο που λέγανε ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι από τη Ρουμανία εργάζονταν στα λιμάνια των κατοχωρών για ένα ευρώ την ώρα ως λιμανεργάτες με μια εταιρεία ταχυδρομική θηρίδα ε, στην ε, Ρουμανία. Και αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Οι Ρουμάνοι εργαζόμενοι δεν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι. Όμω αυτοί που ψάχνουν παραθυράκια στην νομοθεσία δεν θα έπρεπε να μπορούν να τα βρίσκουν. Ήμασταν πολύ βιαστικοί, ήμασταν προθήστε, ήμασταν μάλλον ε, προπετήσε στην αναθεώρηση και την ανανέωση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. είδαμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν μαζί 28 εθνικές αγορές, αρκεί όμως να υπάρχουν τα έχει για την αξιοπρεπή και νόμιμη κυκλοφορία των εργαζομένων και βεβαίως όχι μόνο για την ε, μονόδρομη μετακίνησή τους προς μία κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν να παραδεχτώ ότι η για την απόσπαση των εργαζομένων είναι να βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να υπάρχει μεγαλύτερη κατανομή και ευρύτερη κατανομή των ευθυνών για την απόσπαση των εργαζομένων και όταν αποσπώνται βεβαίως να υπάρχουν οι μισθοί και αμοιβέ. Όμω δεν είναι αυτό το τέλο τη ιστορία. Υπάρχουν ακόμη πολλέ ανισότητε και διαφορέ ω προ τα κοινωνικά επιδόματα και τα πριν που μπορεί να δίνουν τα κάτι μέλη. ό,τι αφορά του Ρουμάνου που εργάζονταν λόγω χάρη στα λιμάνια στι κάτω χώρε, στου λιμένε τη χώρα μου. Ε, το, το ονομάζουμε bonus ή premium shopping στα Ολλανδικά. Να ένα παραθυράκι που έχει αφήσει η νομοθεσία και ε, υπάρχει πολύ περιθώριο για να συνεχιστεί κάτι τέτοιο μέσα από την κοινωνική μας νομοθεσία. Θα πρέπει να προσέξουμε γιατί οι μισθοί πρέπει όντω να είναι ίσοι, οι αμοιβέ να είναι ισότιμες και να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όλοι οι εργαζόμενοι. Έτσι θα διατηρήσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Ευχαριστούμε. Ζλωτόφσκι για ένα λεπτό. Δεν δουλεύει. Α, δουλεύει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ευνηδιάζει λιγάκι τη στιγμή αυτή που διαλέγει για να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα, ε, μια τέτοια μάχη τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε μια τόσο οξία κρίση. Ο περιορισμό τη ε, ελεύθερη κυκλοφορία θα είναι ακριβώ το αποτέλεσμα τη αναθεώρησης τη οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Αυτό προκαλεί την αύξηση τη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίω με την τόσο μεγάλη αύξηση τη ανεργία στην Ευρώπη. Οι καταναλωτέ είναι οι πρώτοι που του απασχολεί αυτό το φαινόμενο. Αυτή θα είναι τα πρώτα θύματα των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ποιο όμω ε, εποφελείται, Ποιο χαίρεται από την... με την πρόταση αυτή. Ακριβώς αυτοί που έχουν το κεφάλαιο στα χέρια τους, οι καπιταλιστές. Αυτό το βλέπουμε διαρκώ στην Ευρώπη που γίνεται όλο ένα και περισσότερο ένα φεουδαρχικό κράτος. Δεν μπορούμε διαρκώ να επιβαρύνουμε τις φτωχότερε χώρες δημιουργώντα κοινωνικέ ανισότητες και βάρη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι έτσι δημιουργούμε ένα σαφή διχασμό μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, ενώ αυτό θέλουμε να το καλύψουμε ω χάσμα. Ευχαριστούμε, κυρία Χάρκιν, για να μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτέλου, έχουμε μια πρόταση αναθεώρηση για την οδηγία απόσπαση των εργαζομένων. Ο Πρόεδρο Γιούνκερ και εσεί η ίδια, κυρία Επιτροπέ, είχατε ε, κάνει δύο φορέ την ίδια προσπάθεια ε, και είχατε πει τα ίδια πράγματα στο ίδιο μέρο. Ε, εδώ σε αυτό την αίθουσα για τον ίδιο σκοπό. Ε, η οδηγία είναι 20 χρόνια, 20 χρονών και είχαμε τόσες υποθέσεις ε, εντωμεταξύ στο ΔΕΚ. Την υπόθεση Λαβάλ μεταξύ άλλων και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Εγώ πιστεύω ότι η αναθεωρημένη οδηγία μπορεί να αντιμετωπίσει πολλέ από τις περιπτώσεις που δημιούργησαν πρόβλημα σήμερα. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα μεταξύ του άρθρου 45 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίση μεταχείριση και του άρθρου 56 που μιλάει για το δικαίωμα των εργαζομένων να παρέχουν υπηρεσίες διασυνοριακά. Το άρθρο 45 διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, για τους εποχιακού και τους προσωρινούς εργαζομένους, για τους μόνιμους ημερικού ε, μερικού χρόνου και για τις ε, γυναίκες. Ε, αλλά όχι για τους αποσπασμένους. Σε κάποιου τομείς, όπως ο κατασκευαστικό, υπάρχουν χάσματα με μεταξύ που φτάνουν το 20% για τις αμοιβέ των αλλοδαπών και εγχώριων εργαζομένων. Και είναι, υπάρχουν χώρε που είναι τεράστιο το μερίδιο το που εκπροσωπούν οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα. Και οι τάσει είναι σε προ τα κάτω των μισθών. Βεβαίω πρέπει να διευκολύνουμε τι επιχειρήσει επιχειρήσει, όπω είπατε και εσεί όμω, ε, Επιτροπέ, ίδια, θα πρέπει να βασιστούμε σε πολλά διαφορετικά κριτήρια. Όχι μόνο στην παραγωγικότητα, αλλά και στην εμπειρογνωμοσύνη, την κοινοτομία, το είδο παροχή ε, που προσφέρεται και όχι αποκλειστικά στου μισθού. Εγώ, όπω του κύριο Κάζα, κύριε Επιτροπέ, σα ευχαριστώ για την τόλμη σα που κάνατε αυτή την πρόταση. Είναι πραγματικά μια καλή αρχή. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λεϊαρίκ για ένα λεπτό. Η δικαιοσύνη και η δημιουργία ενός κοινού χώρου για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους δεν χρειάζεται μια υποτιθέμενη τροπολογία για την απόσπαση των εργαζομένων. Αυτό που προτείνεται διατηρεί την ανταγωνισμό των μεταξύ εργαζομένων εντός της Ένωσης. Θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε μια νέα οδηγία με βάση τη διαβούλευση των συνδικαλιστικών οργανώσεων με στόχο να εξασφαλίσουμε στους αποσπασμένους εργαζόμενους την πραγματική ισότητα μεταχείρισης για τις αμοιβέ, την κοινωνική πρόνοια και τις συνθήκες εργασίας. Θα έπρεπε να συμπληρωθεί από μια συμφωνία για την επιθεώρηση εργασίας ώστε να ε, εφαρμοστεί ένα υψηλό επίπεδο του δικαίου, εργατικού δικαίου Κοινωνικοδημοκρατικέ ε, διαδικασίες για όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενε. Χωρίς αυτό θα απορρίπτεται όλο ένα και περισσότερο αυτέ οι προτάσεις όπως και τώρα. Κυρία Ράιντκε, ένα λεπτό. Uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ, τι επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλείται. Πολλοί πολίτες δεν είναι πλέον πεπισμένοι ότι η Ένωση μπορεί πραγματικά να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις που έχει δώσει και κάποιες φορές ακόμα και εγώ αναρωτιέμαι, κάνουμε αρκετά για να δημιουργήσουμε δίκαιη αγορά εργασίας που προστατεύει τους εργαζόμενους από την εκμετάλλευση, που καθιστά την κοινωνία μας πιο δίκαιη και που να αντέχει τις κρίσεις. Με αυτή την πρόταση για την απόσπαση των εργαζόμενων εργαζομένων ε, μπορούμε να πούμε σαφώς πως δεν πάμε αρκετά μακριά, δεν αποδίδουμε στην υπόσχεσή μας να προστατέψουμε τους εργαζόμενους από την εκμετάλλευση, ειδικά αυτούς που εξαρτώνται κυρίως από μια κοινωνικώς ε, ε, σταθερή νομοθεσία για την απόσπαση. Ε, θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων που διασχίζουν τα σύνορα και, αυτό, και έτσι πολύ συχνά γίνονται πιο ευάλωτοι και χρειάζεται τα κράτη-μέλη να αναλάβουν την επιβολή τη ισχύουσα νομοθεσία. σε σοβαρά. Είναι κρίμα που ζούμε σε μία από τι πιο πλούσιε περιοχέ του κόσμου και δεν μπορούμε ακόμα να προστατέψουμε του εργαζόμενου από παράνομε και επικίνδυνε συνθήκε εργασία από Εργοδότε οι οποίοι χρησιμοποιούν το σύστημα. Ελπίζω πως με μετά από αυτή την πρόταση θα προχωρήσουμε κι άλλο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ατζέα, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκδώσει μια ε, οδηγία εφαρμοστική που έπρεπε να εμποδίσει το κοινωνικό dumping ε, και το dumping των εργαζομένων που έχουν για προς στιγμή σταλεί σε άλλο κατημέλη για να καλυφθούν οι, οι απάτες που έγιναν από αυτές τις ε, εταιρείες βιτρίνες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να κάνει μια σειρά, μια σοβαρή μάλλον ε, πρόταση ε, ωστόσο η οδηγία αυτή αφήνει πολλά κενά γιατί τα κατημέλια έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για να εφαρμόσουν ή όχι του ελέγχου αλλά και τι κυρώσει για να τιμωρήσουν τις ε, περιπτώσεις ε, κατάχρησης. Επιπλέον δίνεται μεγάλη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα και στη βούληση των κρατών μελών να προσφέρουν αυτή τη βοήθεια, αυτή την ενημέρωση στα κράτη υποδοχή ώστε να τιμωρηθούν οι αντικανονικότητες και οι απάτε. Και επίση υπάρχει μεγάλη σύγχυση για την αρχή τη της αναλογικότητας και αυτό θα προκαλέσει και θα αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα αυτής της οδηγίας. Πολλά πράγματα πρέπει να τα συζητήσουμε πλήρως ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Σούλτσε. Κυρία Πίτροπε, κυρία Τάισεν, θέλω να σα ευχαριστήσω καταρχά για τι προτάσει που μα παρουσιάσατε σήμερα και τι λοιπέ τοποθετήσει. Νομίζω αποτελούν μια πολύ καλή βάση με την οποία μπορούμε να εργαστούμε. Είναι σημαντικό, πιστεύω, και στην Ευρώπη να ασχοληθούμε για άλλη μια φορά με το θέμα αυτό και είναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα δεν πάνε όπω θέλαμε σε αυτό το θέμα στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην κατακαιρματίσουμε τις ε, προτάσεις, πρέπει να κοιτάξουμε δεδομένα και με ε, λόγο γνώση. Δεν είναι ο κάθε αποσπασμένο θύμα καταχρήσεων στην Ευρώπη. Πρέπει να κοιτάξουμε βέβαια και την απόσπαση από χώρε ε, χαμηλών μισθών προ χώρε υψηλών μισθών όπου μπορεί να υπάρχουν καταχρήσει, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα ποσοστό 50 με 60% των αποσπασμένων που τίνει προ την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή από χώρε υψηλή μισθολογία σε χαμηλότερου μισθού. Ε, αυτό λοιπόν πρέπει να το κοιτάξουμε. Είτε πρόκειται για το οικοδομικό κλάδο, είτε πρόκειται για σφαγεία και άλλους τομείς. Υπάρχουν πολλές καταχρήσεις που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Εμεί ω Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουμε ζητήσει μια στοχευμένη αναθεώρηση, αλλά πάνω απ' όλα έχει σημασία το περιεχόμενο των όσων περιουλάβουμε σε αυτήν. Και κάτι ακόμα που θέλω να θίξω είναι το ζήτημα τη ίση εργασία, ίσου μισθού στον ίδιο τόπο. Πολύ ωραία ακούγεται αλλά είναι πολύ δύσκολο για να μπω αδύνατο να υλοποιηθεί. Και πρέπει να κοιτάξουμε τι σημαίνει ίσως μισθός, μικτός, καθαρός, ε, ίση εργασία, πώς συγκρίνεται, ίδιος τόπος, ε, κράτη, ίδιο κράτος, ε, ε, περιφέρεια, με ποιο κριτήριο θα προχωρήσουμε, όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ένα λεπτό και τριάντα, Ούλουφσκοπ. Επίτροπε, και εσείς και ο πρόεδρος Γιούνκερ έχετε εκπονήσει μια πρόταση που υποτίθεται ότι θα εξασφαλίσει ίση αμοιβή για παρόμοια δουλειά. Λέτε ότι προσπίσεστε τον κοινωνικό διάλογο και ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι ενώσεις των εργαδοτών θα πρέπει μεταξύ τους να αποφασίσουν το ύψος των αμοιβών και όχι η πολιτική εκ των προτέρων. Αυτό όμως που τώρα πρόκειται να εγκρίνουμε είναι μια πρόταση που ακριβώς πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση. Ε, Άλλα λέγαμε στο παρελθόν με τι διαφορετικέ μα προτάσει. Αυτό που έχουμε πολύ καλά, που έχουμε μπροστά μα, εξυπηρετεί ακριβώ αυτόν τον σκοπό και πρέπει να το εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή. Ε, ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί περισσότερη κινητικότητα ω χώρο εργασία. Ξέρουμε ναι. επίση ότι θα χρειαστούν ίσε αμοιβέ για ίση εργασία. Ναι. Αλλά, ε, κυρία Τάισον, λέτε για μισθούς βιολογικούς, για γυναικείους μισθούς μάλιστα. Μα αυτή είναι αυτομάτως ε, χαμηλότερη από τους μισθούς των ανδρών. Και μετά ε, να συμφωνείτε με τους γεωγραφικώς αιτιολογημένους μισθούς. Πώς γίνεται αυτό. Δεν μου φαίνεται ε, συνεπές. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε στην όλη κατάσταση και θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα σωστής επαναδιατύπωσης της οδηγίας. Η Επιτροπή Απασχόλησης συνεργαστεί στενά μαζί σας για αυτό το σκοπό. Ευχαριστούμε κυρία Λόπες για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν 20 χρόνια τα συνδικάτα ζητούσαν μια οδηγία για να εγγυηθούν την ε, προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων και τότε ε, ε, ξεκίνησε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθέτησε πάνω από τα εργατικά δικαιώματα τα δικαιώματα των εργοδοτών και πρόκειται για μείωση των μισθών υπέρ των κερδών των ε, εργοδοτών. Είμαστε πολύ μακριά από την υπόσχεση του Γιούγκερ που ήταν ίσως μισθός για την ίδια εργασία σε οποιοδήποτε χώρο. Το ίδιο γίνεται και με αυτή την οδηγία. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να είναι εκτός των ε, τομεακών συμφωνιών και πρέπει να περιμένουν 24 μήνες μέχρι ότου εφαρμοστεί πλήρω η εργατική νομοθεσία και στους ίδιου. Εμεί είμαστε αντίθετοι σε μια μήνυμο νομοθεσία που παγιώνει μια προστάτευτη εργατική ε, δύναμη, ενώ έχει αυξηθεί 45% η κινητικότητα αναγκαστικά λόγω της κατάρρευσης των συνθήκων εργασίας από την αρχή της κρίσης. Χρειαζόμαστε μια βαθιά εργατική εναρμόνιση. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτέλου, η Κομισιόν μιλάει για κοινωνική Ευρώπη. Αν και είναι μετριοπαθή αυτή η πρόταση, κάνετε κάποιε χρήσιμε βελτιώσει, όπω α πούμε εγγύηση ίδιο μισθό για την ίδια εργασία στον ίδιο χώρο εργασία, αλλά προσοχή, όχι άλλα συνθήματα. Πρέπει να πάμε πιο μακριά, πιο γρήγορα, με πραγματικέ δικλείδε ασφαλεία, απέναντι στι καταχρήσει τη απόσπαση. Ε, μαύρη λίστα για τι ε, επιτερίες ε, που κάνουν απάτες. Όλα αυτά είναι κρίσιμα πριν να είναι πολύ αργά, κύριε Επίτροπη. γιατί το λέω αυτό. Επειδή το κοινωνικό dumping είναι το σύμβολο της, του αγώνα ανάμεσα στα, σε όσους στην Ευρώπη προστατεύουν και όσους ε, καταστρέφουν. Θα πρέπει να δημιουργηθούν μέτρα πραγματικά προς μια κοινωνική εναρμόνιση προς τα πάνω. Διαφορετικά δικηβεύεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό εμείς οι οικολόγοι αγωνιζόμαστε για μια ευρωπαϊκή ε, ε, επιθεώρηση εργασίας αλλά και για μήνυμο με ευρωπαϊκούς μισθούς, μια ασφάλιση για, την, ε, το επίδομα ανεργίας και μια βιώσιμη ένωση θα έχει αυτό το τίμημα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λένας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει ανάμεσα στα κράτη-μέλη και μέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο όσον αφορά την οδηγία αυτή. Και εγώ πραγματικά συγχαίρω την κυρία Τάισεν που επιμένει για αυτό το θέμα. Είναι μια πρόταση κατά του αθέμητου ανταγωνισμού στην αγορά εργασία. Είναι πολύ σημαντικό και είναι κεντρική σημασία. Πρέπει να είναι δίκαιη όχι μόνο η ελεύθερη ε, κυκλοφορία, αλλά και δίκαιη κυκλοφορία των εργαζομένων. Εμείς ε, θεωρούμε πως η πρόταση ανταποκρίνεται σε δύο βασικές μας απαιτήσει. Καταρχήν η διάρκεια. Πρέπει να είναι προσωρινή απόσπαση και θα πρέπει από αυτές τις βάσεις να ρυθμίζεται. Πώς, ε, ποια είναι η περίοδος ε, βέβαια απόσπασης θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά η πρόταση για περιορισμό της διάρκειας είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αμοιβέ θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, όντω και είναι καλύτερο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο και για την αργόρα εργασία. Πιστεύω ότι ορισμένε προτάσει λοιπόν εδώ είναι πολύ καλέ, είναι ισορροπημένη η πρόταση τη Επιτρόπου Τάισεν και σημαίνει ότι μπορούμε εδώ στο Κοινοβούλιο να αρχίσουμε να την επεξεργαζόμαστε και σωστό να ε, μπορούμε να βρούμε την ισορροπία που χρειάζεται. Σάιμον, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινούσα εξηγούσα στους, εξηγώντας συναδέλφους του UKIP ποιο είναι το όλο θέμα. Ε, και εδώ αυτό που μας απασχολεί είναι να προλάβουμε τις καταχρήσεις της ελεύθερης κινητικότητας των εργαζομένων με σωστές εργασιακές συνθήκες Δεν χρειάζεται τα πράγματα να πάνε Μπορού, θα το εξηγούσα, αλλά δεν βρίσκονται εδώ. Ε, πηγαίνουν ε, να βγάλουν την ομιλία του για να γραφτεί στο YouTube για 60 δευτερόλεπτα και μετά τρέχουν στον μπαρ. Τέλο πάντων, στα 30 δευτερόλεπτα που μου μένουν, να συγχαρώ την Επίτροπο γιατί πραγματικά άκουσε ε, το τι είπαμε και θέλει κάτι να αλλάξει πραγματικά. Ακούσαμε να, λέμε από τους να λένε οι συνάδελφοι πόση ακόμη δουλειά χρειάζεται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα βέβαια στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ίδιο σύστημα. Έχουμε συλλογικές συμβάσεις σε εταιρικό και τομεακό επίπεδο και δεν έχουμε το διάστημα των 24 μηνών, αλλά των 6. Θα φροντίσουμε να παρέχουμε διαφορετική πρόταση, όπως χρειαστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρέγνερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, εξότιμη κυρία Επιτροπή. Είπατε και εσείς η ίδια ότι ο ανταγωνισμός που λαμβάνει η χώρα είναι αθέμητος, μερικές φορές ε, υποβιβάζει τους μισθούς, ε, το κόστος διαβίωσης και εργασίας, δεν προσφέρει δηλαδή όλα αυτά τα υπέροχα και την καινοτομία για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, με την πρόταση που είναι πάρα πολύ σημαντική και που θεωρώ ότι είναι καλή για το ότι επιτέλους έχει καταδεχθεί θέλω να σας απευθύνω μια συγκεκριμένη ερώτηση στην Αυστρία. Ε, ανατίθενται συμβάσεις σε επιχειρήσεις που είναι τελικά οι πιο φθηνές, οι μειοδότες δηλαδή. Και είναι μειοδότες γιατί ε, εργάζονται με απεσπασμένους εργαζόμενους για περίοδο μέχρι δύο ετών. Άρα δεν ε, εισφάλουν, δεν εισφέρουν στο κοινωνικό σύστημα στη χώρα υποδοχής αλλά στη χώρα προελεύσεως δεν έχουν μια καλή συνεργασία οι επιχειρήσεις αυτές διασυνοριακά όπως θέλουμε και ρωτώ εάν οι προτάσεις αυτές τις οποίες ε, καταθέτεται έχουν να κάνουν και με την κοινωνική ασφάλιση και όχι μόνο με την απόσπαση και τη μισθολογική ε, επιλογή. Κύριε Μπενιφέη, ένα λεπτό. Ο κύριος Μπενιφέη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, επιτέλους έχουμε το κείμενο της, τόσο, ε, της ε, οδηγίας που τόσο πολύ περιμέναμε για την απόσπαση των εργαζομένων. Την οδηγία αυτή, όπως και η Επιτροπός Θέσεων, λειτουργεί σε τρία βασικά μέτωπα. Τις αμοιβές των αποσπασμένων εργαζομένων, ακόμα και στην περίπτωση των, ε, ε, της εκμήτρωσης, αποσπάσεις μακρού, μακρού χρόνου και στην κινητικότητα. Θα πρέπει να δούμε το εύρο των διατάξεων αυτών βεβαίω, επαληθεύοντα το αν λίγε τροπολογίε και αλλαγέ που προτείνονται στην πραγματικότητα επιτρέπουν πραγματικά να επιτύχουμε τον επιδιωκόμενο σκοπό. Αυτό που έχει ανακοινωθεί. Δηλαδή ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο. Αυτό είναι η βασική τη της ομάδας μας. Πρώτα απ' όλα η αντίδρασή μου εν θερμό είναι λίγο ανάμεκτη, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να αναθεωρηθεί η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, ενώ όλοι σε αυτή την αίθουσα περιμένουμε ακόμα τα, τη μελέτη τύπου για τι συνέπειε από την αρχή εφαρμογή τη οδηγία αυτή το 2014. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε μια επαρκή θεώρηση του όλου προβλήματο και του φαινομένου και ελπίζω ότι ω Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το κείμενο από κοινού με πλέον συνεργασία. Ευχαριστούμε και τώρα περνάμε στη διαδικασία Και θα να πω ότι από την πλευρά του ΕΛ και μόνο έχουν εγγραφεί έξι αγορητές. Για τις υπόλοιπες ομάδες έχουμε ακόμη μερικούς συναδέλφους. Θα σας έλεγα όμως, επειδή έχουμε καθυστερήσει, να δώσουμε το λόγο σε τρεις συναδέλφους του ΕΛΚ. Και μετά έστω και στους υπόλοιπους. Στους υπόλοιπους που έχουν εγγραφεί. Φάντερ Κέλλερε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι. Καμία πρόταση δεν είναι τέλεια. Ακόμη και αυτή που υποβλήθηκε από την Επίτροπο Τάισεν δεν θα είναι τέλεια. Για κάποιους ε, ξεπερνάει τα όρια, για κάποιους είναι επαρκής. Ωστόσο, η πρόταση είναι ισόρροπη. Αυτή είναι η αξία της. Ε, εδώ δίνεται τουλάχιστον κάποια προσοχή στα δικαιώματα των εργαζομένων και δημιουργούνται κάποιοι κανόνε για τι επιχειρήσει αλλά και κάποια διευκόλυνση στο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η Επιτροπή στα περιθώρια που έχει. Βασίζεται τουλάχιστον στην αρχή ίση εργασία, ίσε αμοιβέ μάλλον για ίση εργασία στον ίδιο τόπο. Και αυτό αξίζει την αναγνώρισή μα και τι ευχαριστίε μα. Η Επιτροπή με την πρόταση αυτή δίνει το καλό παράδειγμα. Εμεί ω βουλευτέ και θα πρέπει να φροντίσουμε να να βελτιώσουμε την κατάσταση για να αποφύγουμε προφανώς να υπάρξουν περαιτέρω παραβιάσεις σε επίπεδο κατομελών. Ξέρουμε ότι η ψηφιακή συνεργασία μεταξύ των κατομελών είναι η μόνη πραγματική εγγύηση που θα επιτρέψει να ε, ξεπεράσουμε τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργεί αυτή η κατάσταση. Και αυτό μπορεί να γίνει αρκεί να υπάρχει διάθεση, αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προ του ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστούμε. Ο κ. Επίτροπε, η προσπάθεια που έκανε η Επιτροπή είναι σίγουρα χρήσιμη. Το αποτέλεσμα όμως απογοητευτικό. Εγώ βλέπετε δεν έχω καμιά αντίρρηση στην ελεύθερη κυκλοφορία. Αντίθετα πιστεύω πως η κινητικότητα μπορεί να είναι ένα σημαντικό μέσο στα ανταγωνιστικά μοντέλα, στα συστήματα επιχείρησης και στις εταιρείε. Όμως ε, θα πρέπει να υπάρχει ισότητα ε, ε, ρυθμίσεων, κανόνων, αμοιβών και κοινωνικής πρόνοιας. Διαφορετικά η μετακίνηση σημαίνει κοινωνικό dumping και εργασιακό dumping για όλους τους ανθρώπους που ε, εμπλέκονται. Η ισότητα στην πρόταση που κάνατε δεν υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναρχίσετε αυτό και από την αρχή. Και θα πρέπει να το κάνετε με μεγάλη προσοχή, γιατί εντωμεταξύ η κατάσταση δεν μένει σταθερή. Και θέλω να πω δύο πολύ σύντομα πράγματα σε σχέση με το χρόνο για τη σταθεροποίηση. 24 μήνε δεν είναι μόνο πολύ. Είναι και αντίθετα με αυτό που προβλέπετε, για παράδειγμα, στην οδηγία για την εποχική, εποχική εργασία. Επίση, θα ήθελα να θυμίσω σε όλου ότι στη συμφωνία που έγινε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν, υπάρχουν κανόνε που αλλάζουν την προστασία των ατόμων. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, η οδηγία πραγματικά συμβάλλει στο να μην έχουμε κοινωνικό ντάμπινγκ κατά των εργαζομένων, στο να μπορούμε να έχουμε κινητικότητα των εργαζομένων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμω υπάρχει μια διγλωσία και η διγλωσία είναι η εξή. Στη συμφωνία που έκαναν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων για τη διευθέτηση του ζητήματος της Βρετανίας υπάρχουν πλέον διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες θα υπάρχει διακριτική μεταχείριση για λόγους ηθαγένειας όσων νεοεισερχόμενων εργαζομένων στην αγορά εργασίας της βρετανίας και δεν θα έχουν δικαιώματα που πηγάζουν από τις εργασιακές σχέσεις δεν θα έχουν επίδομα κατοικίας δεν θα έχουν φοροαπαλλαγές δεν θα έχουν άλλα επιδόματα. έχει σχέση αυτό άραγε με την ευρωπαϊκή ένωση; τι συζητούμε. γίνεται διάκριση εις βάρος των εργαζομένων για λόγους ηθαγένειας. αυτό είναι εις βάρος 400.000 ελλήνων επιστημόνων. το ίδιο και για άλλους. Πώς μιλούμε λοιπόν εδώ για κινητικότητα των εργαζομένων. Να σταματήσει η διγλωσία επιτέλους σε αυτό εδώ το σώμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η μανία των ε, κρατών μελών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να πάρουν μεγαλύτερες ποσοστώσεις στην οικονομία ενώ αφήνουν κατά μέρο την πιο σημαντική σύγκληση, την κοινωνική σύγκληση ενώ οι ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών περνούν από μια Ευρώπη πραγματικά κοινωνική δεν μπορούμε να κάνουμε ε, τους σκοφούς και να κοιτάμε από την άλλη μεριά. Θα πρέπει να φτιάξουμε μια Ευρώπη με ίσια δικαιώματα, κοιτώντας προς τις πιο δημοκρατικές και τις πιο αναπτυγμένες κοινωνικά χώρες. Χρειαζόμαστε μια, ένα διοικητικό μηχανισμό που θα οδηγεί σε μείωση των ανισοτήτων. Όσο λειτουργούμε με συμμετρικό τρόπο, στην ουσία δεν ανταποκρινόμαστε στι ευρωπαϊκέ αξίε. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν στόχο να σταματήσουν το κοινωνικό ντάμινγκ θα πρέπει να στηριχθούν. Στηρίζουμε την αναθεώρηση τη οδηγία για του αποσπασμένου εργαζόμενου και εργαζόμενου που πραγματικά θα καλύπτει τα κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα για όσου εργάζονται εκτό των συνόρων του και θα καταπολεμά τι ε, μη θεμητέ πρακτικέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η κυρία Μόρα Σαχτιέ Ξεκινώντας και προτείνοντας αυτή την οδηγία, ξεκινάτε μια έναν αγώνα κατά των λαϊκιστών που θέλουν να τονίζουν την εθνικιστική αναδίπλωση. Είστε πολύ θεραλέα. Χρειάζεται όντως περισσότερη κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να διευκολύνουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη δυναμική των επιχειρήσεων και όλοι εδώ να έχουν δουλειά και κοινωνική προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, εργαζόμαστε μέσω αυτού του κειμένου για όλους τους Ευρωπαίους εργαζόμενους για τη δυναμική της απασχόλησης και οφείλουμε να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη ώστε να καταπολεμήσουμε την απάτη, να εφαρμόσουμε αυτά τα ευρωπαϊκά κείμενα για να οικοδομήσουμε εδώ όλοι από κοινού και άκουσα πολύ προσεκτικά τα σημεία συνένεση τα οποία μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε όλοι μαζί, να γνωρίζετε κύριε Επίτροπε ότι εμεί θα είμαστε στο πλευρό σα. Ευχαριστώ. Κυρία Ρουόνεν, από την ECR ζήτησε το λόγο και επειδή λείπει ένα συνάδελφο από το ΕΛΚΑΡ, πιστεύω ότι μπορούμε να τη δώσουμε το λόγο. E Σας ευχαριστώ. πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναζητούν εργασία σε άλλες χώρες εκτός της δικής τους, είναι οι περισσότεροι πολύ μορφωμένοι και επιπλέον υπάρχουν και, άλλο 1,5 εκατομμύριο διασυνοριακοί εργαζόμενοι. Υπάρχουν και αποσπασμένοι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν σύντομες ε, συμβάσει για εργασία εκτός της χώρας τους. Άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο κόσμος Εν πάση περιπτώσει, όποια ομάδα και αν εμπίπτει, αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχει την ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία. Δεν θα πρέπει να έχουμε αγορά εργασία δύο επιπέδων, όπου οι ξένοι, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι θα πληρώνονται λιγότερα χρήματα από του ε, ηθαγενείς. Ε, αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και είναι για αντίθετο στις θεμελιώδεις μας αξίες. Ευχαριστώ πολύ. Σόγκορ Τσάμπα. Συμφωνώ με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ανάπτυξη οποιασδήποτε νομοθεσία θα πρέπει να βασίζεται σε ενήμερη απόφαση. Και γι' αυτό δεν βλέπω τη λογική της τροποποίησης αυτής της οδηγίας πριν να, έχει ε, ε, εφαρμοστεί η η οδηγία για την εφαρμογή και πριν να έχουν γίνει αισθητά τα επιτελέσματά της. Νέα δράση θα πρέπει να γίνει όταν και αν φανεί πως αυτή η οδηγία δεν αρκεί. Κυρίως σε αυτή την περίπτωση όπου μιλάμε για βασικές αρχές της, ε, ε, της ε, κοινή αγοράς, ελεύθερη κυκλοφορία, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε στις προσπάθειές μας καταπολέμησης, κατάχρησης και απάτης που συμφωνώ ότι χρειάζονται να μην διατρέξουμε τον κίνδυνο να δημιουργήσουμε νέους φραγμούς για την κινητικότητα των εργαζομένων και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. ευχαριστώ πρόεδρε ευχαριστώ το σώμα για αυτή την τόσο ε, συνεπτική συζήτηση και το λέω γιατί και μέλος υπήρξα αλλά είμαι και ευγνώμων για τις τόσες πολλές συνεισφορές των συναδέλφων για κάποιους από τους, βουλευτές η πρόταση δεν είναι αρκετή, για κάποιους είναι υπερβολική. Σίγουρα το θετικό να δεν αφήνει κανένα διάφορο. Και βλέπω ότι είναι αρκετοί εκείνοι μεταξύ των βουλευτών που είναι πρόθυμοι να ακούσουν ο ένας και να σεβαστούν ο ένας τις απόψεις του άλλου. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο για να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Βλέπω πάντως ότι ε, η πρόταση αυτή είναι κάτι που όλοι το επιθυμούν. Και πολλοί με ρωτήσαν γιατί δεν περιμένουμε μέχρι η εφαρμοστική οδηγία να αποτιμηθεί. Αυτή που είχε, το είχε αρχίσει να, λειτουργεί, να ισχύει το 2014 και μετά να προχωρήσουμε. Όμως η εφαρμοστική οδηγία στόχο είχε να παράσχει περισσότερα εργαλεία, περισσότερα μέσα στα κατημέλη για να μπορέσουν να έχουν καλές επιδόσεις στην υλοποίηση. Η εφαρμοστική οδηγία ήδη υπάρχει και λειτουργεί σκοπό έχει να καταπολεμήσει την εξαπάτηση και τις απάτες. Ε, ο σκοπός λοιπόν ήταν να έχουν ένα πιο ε, πλούσιο πλουστάζιο τα κρατη Εδώ τώρα ενθαρρύνουμε τα κρατη να υλοποιήσουν την οδηγία αυτή εγκαίρως με τρόπο αποτελεσματικό προκειμένου να ε, είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πρέπει όμω και οι ίδιοι να δούμε του κανόνε, πώ εφαρμόζονται και πώς υλοποιούνται και να δούμε αν υπάρχουν ανεπάρκειε. Αυτό σα υποσχεθήκαμε και εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μα, ότι θα δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό το θέμα, θα ε, επικεντρωθούμε στην αναθεώρηση, προκειμένου να πετύχουμε την ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο. Αυτό ακριβώ θέλαμε και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να περιμένουμε μέχρι να αποτιμηθεί η εφαρμοστική οδηγία. Τώρα επιτέλου έχουμε και το, την κατάλληλη συγκυρία και την ευκαιρία για να ανταλλάξουμε απόψει για τι τεχνικέ λεπτομέρειε, για τι τεχνικέ λεπτομέρειε που πολλέ φορέ είναι κεφαλιά, Πρέπει να δούμε λόγω χάρη τα έντυπα Α1, τα οποία δείχνουν ή αποδεικνύουν εάν τα κοινωνικά επιδόματα ε, καταβάλλονται, αν οι σφορέ καταβάλλονται σωστά. Γιατί έχουμε και άλλες προτάσεις που τρέχουν παράλληλα για την ε, ευθυγράμμιση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Τα έντυπα λοιπόν αυτού του είδους ε, θα γίνουν πιο αξιόπιστα, πιο ε, αποτελεσματικά και τα κάτι μέλη θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι, όπως είπαμε και πριν και για τη διοργανική συμφωνία, με το νομοθετικό μας πλαίσιο καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε εύληπτη νομοθεσία. Όχι μακροσκελή κείμενα που κοστίζει να τα διαβάσει και μόνο κανείς. Είπαμε να είμαστε απλοί σε επίπεδο επιμέρους εταιριών να ε, εκπονείται η νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε την ίδια κατεύθυνση και σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στις συλλογικές ε, συμφωνίες και να σεβαστούμε τις προτεραιότητες των κοινωνικών εταίρων. Αυτό που επίσης θέλω να τονίσω και να υπογραμμίσω είναι αυτό που είπα και στην ε, εισαγωγική μου ομιλία. Δηλαδή, να πετύχουμε κινητικότητα για όλη την Ευρώπη. Αλλά με σαφείς κανόνες, με δίκαιους κανόνες, με κανόνες που να μπορούν να εφαρμοστούν παρομοίως παντού. Αυτό όμως που χρειαζόμαστε είναι επίσης κανόνες που να τους αποδέχεται το ευρύ κοινό, οι πολίτες. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι, αλλά να γινόμαστε και αντιληπτοί ως δίκαιοι. Πραγματικά ανυπομονώ για τη συνέχεια της συζήτησης και περιμένουμε τις απόψεις των ε, κρατών μελών και των βουλευτών με αδημονία. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που έχουν ε, θετικό ε, πνεύμα συνεργασίας μαζί μας. Πιστεύω και θα μας εξυπηρετήσουν να πετύχουμε όλοι τον κοινό μα στόχο. Ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Κύριε Σταβελό, θέλει κάτι για το ημερήσια διάταξη, παρακαλώ. Πρόεδρε, θα ήθελα επί του κανονισμού να με καθησυχάσετε γιατί πιστώνω ότι αυτή η συζήτηση για την απόσπαση των εργαζομένων λαμβάνει χώρα χωρίς παρουσία κανενός ε, μέλους της άκρας δεξιάς, της ΕΝΕΦ e όπως ονομάζεται, του ε, Εθνικού Μετώπου. Ε, εσείς τους είπατε ότι δεν έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν ή μήπως δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αυτή η συζήτηση. Γιατί είναι κάτι το οποίο σε κάθε εκλογική εκστρατεία μας πίζουν τα αυτιά. Συνέχεια μας μιλούν για, τα, για την Ευρώπη και τα εργασιακά δικαιώματα. Μήπως έπρεπε να είναι παρόντες στη συζήτηση αυτή σήμερα. Καλώς πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης και εδώ έχουμε